Allora, buongiorno a tutti. Καλημέρα σε όλους. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε επειδή έχουμε δύο εισηγήσεις. που θα ήθελα να έχουμε χρόνο αυτό να τη συζητήσουμε πριν περάσουμε στις ψηφοφορίες. Ακόμη λοιπόν και όταν έχουν φτάσει όλοι οι συνάδελφοι, θα έλεγα να περιμένουμε δύο λεπτά και μετά θα ζητήσω από, θα ζητήσω από τον συνάδελφο Κάνφιλντ, Κάλφιν, συγγνώμη, να ξεκινήσει την παρουσίαση της εκθεσής του. Έχουμε στη διάθεσή μας 30 λεπτά για τη συζήτηση αυτή. Και μετά θα συζητήσουμε την έκθεση Γκιουρκ. E Θα έλεγα λοιπόν, αν μπορεί ο συνάδελφο Κάλφιν να μα παρουσιάσει την εκθεσή του για την προστασία των υποδομών πληροφοριών ζωτική σημασία, επιτεύγματα και επόμενα βήματα προ την παγκόσμια ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Παρακαλώ. Thank you uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αυτή είναι μια έκθεση κατά πρωτοβουλία η οποία είναι στενά συνδεδεμένη με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρουσιάστηκε το 2011 και ουσιαστικά αναφερόμαστε εις το θέμα το οποίο για πολλούς λόγους απέδειξε ότι έχουμε την δυνατότητα να συζητήσουμε ε, την σημασία της ασφαλείας στον κυβερνοχώρο και ε, όπως σας είπα η έκθεση αυτή έχει συνδυαστεί με το πρόγραμμα δράσης για την ε, πληροφόρηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα του cloud computing ε, και του διαδικτύου στα σύννεφα αν μπορούμε να το, να, να το εκφράσουμε έτσι και ε, επιπλέον έχουμε ε, το θέμα της προστασίας των δεδομένων ε, υπάρχει στην Επιτροπή μας το θέμα αυτό. Ψηφίσαμε για την ΕΝΙΣΑ και όλες οι εξελίξεις αυτές έχουν στενή σχέση με τη χρήση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών διότι η ανάπτυξη του ίντερνετ πρέπει να μας εξασφαλίζει ότι θα έχουμε ένα ανθεκτικό δίκτυο το οποίο θα επιτρέψει να αναπτύξουμε την ε, νομοθεσία σχετικά με το διαδίκτυο και ε, αντιλαμβάνομαι ότι έχει, υπάρχουν ε, τρεις ομάδες προτάσεων και γι' αυτό πολύ σύντομα θα το εξετάσω. Ο, καταρχάς αναφερόμαστε εις την ε, προστασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ε, θέλουμε να ενισχύσουμε την σχετική νομοθεσία η οποία υπάρχει αλλά έχει πολύ ε, περιορισμένο εύρος και γι' αυτό πρέπει να αλλάξει δομή διότι ε, η υποδομή είναι πολύ περιορισμένη και δεν προσεγγίζει ούτε ε, από μακριά την αμερικανική ε, νομοθεσία σχετικά με το υπερλογιστικό νέφος. Οπότε πρέπει να δούμε ποιες είναι οι τεχνολογίες που περιλαμβάνονται και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε χρησιμοποιήσουμε μηχανισμούς οι οποίοι είναι ήδη κατηρτισμένοι κατά τρόπον ώστε να δημιουργήσουμε ε, μία ανθετική υποδομή για το διαδίκτυο. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν χωρίς την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ ιδιωτών και δημοσίου και ε, χαίρομαι διότι υπάρχει τεχνολογία κατάλληλη και το εξετάζουμε στη δικιά μας επιτροπή διότι κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να υιοθετήσουμε την άποψη της τεχνολογικής εξελίξεως και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Βεβαίως θέλω να συγχαρώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι εκπονεί τις διάφορες στρατηγικές και είναι στη διάθεσή μας για διαβουλεύσεις ε, ε, και ε, για συνεργασία με τους σημαντικότερους παίκτες στο χώρο αυτό. Πρέπει να ενισχύσουμε τη δυνατότητα να ενισχυθούν τα εθνικά προγράμματα για ανταλλαγή κρισίμων πληροφοριών, να έχουμε ε, διάφορους ε, ε, υπευθύνους συνδέσμους, άτομα δηλαδή που να εξασφαλίζουν την συνεργασία μεταξύ των κρατών και στα πλαίσια αυτά και σε σχέση με την εργασία που έχει γίνει στην Επιτροπή σχετικά με την ΕΝΙΣΑ διαπιστώνουμε ότι είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για να προωθηθεί αυτό το σημαντικό θέμα που άπτεται του διαδικτύου. Όσον αφορά την ασφάλεια του διαδικτύου, ουσιαστικά έχουμε μία σειρά προτάσεων που αποβλέπουν στο να υπάρξει ένας καλύτερος συντονισμός μεταξύ των ομάδων αντίδρασης ε, και να ε, ενισχύσει την εργασία την οποία κάνει η ΕΝΙΣΑ εφόσον εξασφαλίσουμε ελάχιστη ε, αντίδραση ε, ελάχιστα ε, πρότυπα ε, σχετικά με τις αντιδράσεις που χρειάζονται για να αντιδράσουμε και να προλάβουμε ενδεχόμενες επιθέσεις στο διαδίκτυο. Αντιλαμβανόμαστε ότι ε, οι χώρες μέλη έχουν διαφορετικό βαθμό εξελίξεως μεταξύ τους, οπότε είναι δύσκολο να έχουμε μία ασφάλεια ελαχίστου επίπεδου που θα καθησυχάσει τους χρήστες του διαδικτύου. Προτείνω λοιπόν στην έκθεση κάτι το οποίο ε, ενδέχεται να προκαλέσει συζητήσεις και εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δηλαδή ε, την ε, κοινοποίηση για μία παραβίαση της ασφαλείας και όποτε δηλαδή υπάρχει μία παραβίαση της ασφαλείας της μεταφοράς πληροφοριών να υπάρχει εγκαίρως μία ειδοποίηση ε, και ε, να ε, εντοπίζεται το πρόβλημα, πράγμα το οποίο θα επιτρέψει στις εταιρείε να έχουν ένα επιπλέον κίνητρο για να δημιουργήσουν τους αναγκαίους μηχανισμούς προστασίας και ασφαλείας ο στόχος μας λοιπόν είναι να υπάρχει μία συνέπεια και συνέχεια σε όλα τα κράτη-μέλη, να ενισχύσουμε τις ε, ε, τις προσπάθειες για την ε, επιμόρφωση και την εκπαίδευση σε όλες τις χώρες στον τομέα αυτό και βλέπουμε ότι ορισμένες χώρες ηγούνται ότι η συνειδητοποίηση του κοινού μπορεί να βοηθήσει να προληφθούν παραβιάσεις ε, της ασφαλείας μεταδόσεως των πληροφοριών και ε, να υπάρχει μία στρατηγική Εσωτερική εσωτερικής διεκπαιρεώσεως της ασφαλείας και η στρατηγική αυτή ε, δεν πρέπει να είναι ένα πρόγραμμα κλιμακωτό αλλά να υπάρξει μία βάση η οποία θα συγκεντρώσει και θα συντονίσει όλες τις προσπάθειες να εξασφαλίσουμε ασφάλεια στο διαδίκτυο με τον ίδιο τρόπο που διεκπαιρεώνεται και στις Ηνωμένε Πολιτείες είναι καλό ότι αυτό εξελίσσεται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και τέλος κύριε Πρόεδρε, έχω λίγα πράγματα να πω ε, σχετικά με ένα βασικό μέρος της εκθέσεως, διότι τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει παρουσιαστεί σωστά εις ε, τους διάφορους οργανισμούς, διότι δεν υπάρχει ο σωστός μηχανισμός και μόνο τα τελευταία ένα-δύο χρόνια έχει προχωρήσει αυτή η εξέλιξη με την ε, προώθηση της ασφαλείας στον κυβερνοχώρο με ε, περισσότερες συντονισμένες ενέργειες ε, για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ενώσεως αλλά υπάρχουν ακόμη πολλά κενά χρειάζεται συνεργασία και σε εθνικό επίπεδο η οποία είναι ε, ε, πιο σταθερή αλλά δεν υπάρχει τόσο καλή συνεργασία διεθνώς. Χρειάζεται λοιπόν οι σχετικοί οργανισμοί να περιλάβουν αυτό το θέμα εις ε, τα πλαίσια της δράσεως της ε, υπηρεσίας εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε συντονισμό με τις Ηνωμένε Πολιτείες με τις οποίες υπάρχουν ειλικρινές και ανοιχτές ε, εμπορικές σχέσεις κατά τρόπον ώστε να εξεταστεί το θέμα από αυτή την οπτική γωνία διότι μόνοι μας ό,τι και να κάνουμε δεν θα υπαρκέσει. Τέλος πρέπει να περιλάβουμε το θέμα αυτό εις ε, τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στα, ε, ε, στους διεθνείς οργανισμούς, στον ΟΣΑ, στο G20 ε, και αυτές είναι οι προτάσεις τις οποίες έχουμε σχετικά με τις τρεις αυτές ενότητες θεμάτων που θα εξετάσει η έκθεση και ε, θα μπορέσουμε να προωθήσουμε ένα συνεκτικό έργο ως όφελος της ε, ασφαλείας στον κυβερνοχώρο. Ευχαριστώ τώρα ο κύριος Βανίστελ Ρόι Σκιώδης, ευχαριστώ Πρόεδρε. Σύντομα θα τα πω σήμερα το πρωί για αυτό το θέμα. Γιατί είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και διαρκή ε, κάθε φορά που χρειαζότανε. Ακριβώς αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ σημαντική όσο και επίκαιρη η έκθεση για να τοποθετηθεί η Επιτροπή μας. Το κοινοβούλιο κάνει σαν να ε, υπάρχει θέμα ιδιωτικής σφαίρας. Κοιτάξτε, ε, στο διαδίκτυο υπάρχουν κάποια θέματα σημαντικά, θέματα ασφαλείας και μέτρα ασφαλείας. Αν κοιτάξετε να δείτε τι γίνεται και πώς αναπτύσσεται η οικονομία μας και τι αναμένεται στο μέλλον, τα πάντα από το online banking, τραπεζικές εναλλαγές κάνουν οι πολίτες από το διαδίκτυο και τόσα άλλα. Ε, είναι σαφέστατο λοιπόν και πεντακάθαρο το είπατε και εσείς στην έκθεσή σας. Από την άλλη, φροντίσατε να μείνετε στο μονοπάτι της Ήτρε και να μην μπείτε σε άλλα χωράφια. α πούμε ασφάλεια ε, πολύ συγκεκριμένων στοιχείων του διαδικτύου που δεν μας αφορούν. Ε, είμαι πολύ ε, θετικός για την έκθεση. Έχω να κάνω τρία σχόλια. Πρώτον, μέχρι πότε θα περιμένουμε τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν. Η μία χώρα λέει η κατάσταση είναι ε, ε, ε, κόκκινος συναγερμός, η άλλη χώρα λέει είναι πορτοκαλί και η άλλη λέει είναι κίτρινο. Τι σημαίνει αυτό τώρα. Ας πούμε ότι υφίσταται επίθεση μια τράπεζα που εξαρτώμαστε τόσο πολύ. Όλες οι χώρες δεν το χαρακτηρίζουν στο ίδιο επίπεδο κινδύνου και ασφαλείας. Και βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει ψηλή ασφάλεια, ε, αλλά να μην είναι κάτι το ειδικό για το Λουξεμβούργο, για τη Δανία, για τη Λιθουανία, α πούμε, φτιαγμένο. Θα πρέπει να υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να μετράει. Και τι μπορούμε ε, να μάθουμε. Πολλά μπορούμε να μάθουμε ε, ο ένα από τον άλλο. Είναι πολλά τα καλά παραδείγματα, αλλά παραμένουν στην περιπτωσιολογία. Εμεί θέλουμε να υπάρχει ασφαλής κυκλοφορία και ασφαλή οικονομική εξέλιξη και στο διαδίκτυο. Κάτι άλλο σημαντικό το συζητήσαμε είναι η σημασία των επιχειρήσεων. Να, όχι μόνο οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις που συνεργάζονται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μάλιστα και σε παγκόσμιο πολλές φορές. Χρειάζεται λοιπόν και το ευρωπαϊκό επίπεδο σε συνεργασία των επιχειρήσεων. Και θα πρέπει να τοποθετηθεί και σε αυτό η Επιτροπή μας στη μελλοντική συζήτηση και θα έλεγα, Πρόεδρε, ότι αυτό δεν θα γίνει αυτόματα εμείς είμαστε η Επιτροπή για το Διαδίκτυο, εμείς είμαστε η Επιτροπή ε, που είναι αρμόδια για όλες τις εξελίξεις στη βιομηχανία και στην τηλεκοινωνία. Λοιπόν, αυτές τις τρεις παρατηρήσεις είχα, είναι εξαιρετική η έκθεση. Θα κάνω κάποιες τροπολογίες, αλλά όχι και τρομερές, γιατί έχουμε συνεργαστεί πολύ καλά μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Thank you very much, Ευχαριστώ πολύ κύριε Βανίστεροι. Ο κύριος Κρόιτσμαν. Θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το θέμα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, στο μεταξύ, ε, το συζητούν όλοι. Και αν διαβάσετε τον τύπο αυτές τις μέρες, οι Αμερικανοί ε, δήλωσαν ότι θα μπορούσε να υπάρξει και επίθεση. Γι' ε, αυτό συνιστά επίθεση κατά της ασφάλειάς τους και θα μπορούσε να απαντηθεί και με στρατιωτικά παρακαλώ μέσα. θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό και να μας απασχολήσει. Έχουμε εξάρτηση σήμερα από υποδομές, ε, επικοινωνίες και ε, οι πολίτες και τα κράτη χρειάζονται συστήματα φερέγγια που δεν ε, επιτρέπεται να καταραίουν σε έκτακτες περιστάσεις. Το λέει και ο εισηγητής η εμπιστοσύνη στις υποδομές μας είναι από τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και την ευημερία. Πολλά επεισόδια τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο στην Ευρώπη έχουν κλονίσει αυτή τη σημαντική εμπιστοσύνη και φάνηκε ότι και κρατικές υπηρεσίες αλλά και επιχειρήσεις χρειάζονται να δράσουν. Στενή συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων, της οικονομίας και των κρατών μελών θα πρέπει να παραμένει προτεραιότητα. Επειδή είναι πολύ μεγάλη δικτύωση στην Ευρώπη, ε, η διασύνδεση θα πρέπει να συνεννοούνται τα κράτη-μέλη και να εκπονήσουν στρατηγικές και προγράμματα έκτακτης ανάγκης για να εντοπίσουν τα αδύνατα σημεία για να τα ε, καλύπτουν από κοινού. Ε, σημαντικό ρόλο καλείται εδώ να παίξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίως θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα έχουμε και την απαραίτητη πραγματογνωμοσύνη. ορίζουμε τις προτάσεις ε, οργανισμός ε, που είναι αρμόδιος στη Ένωση για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, ο ΕΝΙΣΑ, καλό θα ήταν να έχει μεγαλύτερες αρμοδιότητες για να μπορεί να εξασφαλίζει και να εγγυάται μεγαλύτερη ασφάλεια. Ε, και μεγαλύτερη πρόληψη στον προγραμματισμό χρειάζεται. Δηλαδή η χρήση των συστημάτων υπολογιστών, είτε είναι ιδιώτες, είτε είναι φορείς οικονομίας, θα πρέπει να συμμετέχουν. Πρότυπα ασφαλείας θα μπορούσαν εδώ να βοηθήσουν. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να είναι νομικά δεσμευτικά και νομοθετικά. Να το σκεφτούμε. Πολλές φορές οι νομοθέτες και οι κρατικές αρχές υπολείπονται των εξελίξεων. Θα πρέπει λοιπόν να περιορίζονται αυτά τα μέτρα στα ελάχιστα και να ε, είναι προϊόν συνεργασίας με τους ε, παραγωγούς των συστημάτων ε, τηλεπικοινωνιών γιατί έχουν και την πρακτική εμπειρία και την πραγματογνωμοσύνη. είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεργασία αυτή γιατί ένα τεχνικό συμβάν επεισόδιο που προκύπτει σε μια χώρα μπορεί να αφορά και άλλη χώρα. Οι απειλέ δεν γνωρίζουν σύνορα ούτε εθνικά ούτε εξωτερικά τη Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει και διεθνώ να δραστηριοποιηθεί και να φροντίσει για μεγαλύτερη συνεργασία. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή τον κύριο Κάλφιν για την έκθεσή του. Το σχέδιο έκθεση είναι πολύ καλή αφετηρία για συζήτηση και χαίρομαι για τη μελλοντική συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κρόιτσμαν. Δεν ζήτησε άλλο κανεί το λόγο. Η κυρία Γκροστέτ, παρακαλώ. Ε, merci beaucoup. Ε, ευχαριστώ. Εδώ το ζήτημα που μας απασχολεί είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Είδαμε ότι τα θεσμικά όργανα της Ευρώπης δεν μπορούσαν να αποφύγουν τις επιθέσεις κατά των ίδιων των ιστοτόπων τους και γνωρίζουμε σήμερα ότι υπάρχει ένας αριθμός χωρών που ονομάζουμε αναδυόμενες αλλά δεν είναι πια αναδυόμενες όπως η Κίνα που αναπτύσσουν όπλα συγκεκριμένα όπλα, οπότε θα πρέπει να αγωνιστούμε για να αναχαιτήσουμε τον κυβερνοπόλεμο. Κυβερνοπόλεμο τον οποίο θα μπορούσε να διεξάγουν κάποια κράτη όπως η Κίνα αλλά και άλλοι έχουν τα μέσα για να το πραγματοποιήσουν. Η κινέζικη κυβέρνηση δεν αγνοεί τις δυνατότητες που τους προσφέρουν τα νέα αυτά τεχνολογικά μέσα και πέραν της λογοκρισίας που ισχύει εντός της χώρας εκμεταλλεύεται τις ε, δυνατότητε των δικών μα δικτύων για να έχει το μέγιστο των πληροφοριών και να μα αποδυναμώσει έστω και προσωρινά. Στι αρχέ του 2011, οι κινέζικε αρχέ δήλωναν ότι δημιούργησαν μια υπηρεσία κύβερνο άμυνα. Οπότε συνειδητοποιούμε ότι είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασχοληθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με το όλο ζήτημα. Θα πρέπει να καταφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, δει συνδυαστικά όσα συμβαίνουν στο κάθε κάτω μέλο. Διότι το ερώτημα είναι, είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε κατά των νέων αυτών απειλών στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε τι δυνατότητε και τι τεχνολογικέ και τι ε, οργανωτικέ. Αυτά ήθελα να πω. Έδωσα το παράδειγμα τη Κίνα απλώ, αλλά είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν και άλλα. Ε, εδώ δεν θα πρέπει να είμαστε αφελείς ω προ το συγκεκριμένο ζήτημα. Κάποιε φορέ τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα υπήρξαν ιδιαίτερα αφελή. Όχι. Θα πρέπει να προβλέψουμε το τι ε, πρέπει να γίνει κατά πρώτον, συνδυάζοντα τα όσα γίνονται στα διάφορα κράτη-μέλη και προσπαθώντα να έχουμε μια ευρωπαϊκή μορφή προστασία. Ο κύριος Ανέν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε το διαδίκτυο έχει γίνει ένα καθοριστικό στοιχείο τη καθημερινή ζωή πολλών Ευρωπαίων πολιτών. Από το διαδίκτυο μπορεί κανεί να κλείσει ένα δωμάτιο σε ξενοδοχείο, να λύσει τα τραπεζικά του προβλήματα, να παραγγείλει, να αγοράσει, να πωλήσει, να επικοινωνήσει, να δώσει πληροφορίε λίγο πολύ ε, μυστικές, απόρριτες, προσωπικές. Είναι λοιπόν ε, ένα απόσπαστο στοιχείο της καθημερινότητας των πολιτών και της οικονομίας. Έχω την αίσθηση ότι στην όλη αυτή υπόθεση ε, παραλαμβάνουμε τα λάθη που είχαν γίνει και στο παρελθόν όταν δημιουργήσαμε την Ιντερπόλ και έπρεπε να έχουμε ένα είδο αλληλεγγύη ώστε να καταφέρουμε ομαδικά να αντιμετωπίσουμε την εγκληματικότητα. Σήμερα για το διαδίκτυο είναι προφανέ ότι όσοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο για να επιτεθούν σε άλλου είναι πιο μπροστά σε σχέση με την ε, δική μας την αντίληψη του θέματος. Γι' αυτό λοιπόν η έκθεση έχει, θα έπρεπε να έχει περισσότερο συνολική θεώρηση, να παρουσιάζει περισσότερο συνολικά μέσα για να προστατεύσει του Ευρωπαίου πολίτε από επιθέσει που θα μπορούσαν να προκύψουν και σήμερα ακόμη. Πολιτικέ επιθέσει ή και εγκληματικέ. Θα πρέπει λοιπόν να δράσουμε με ταχύτητα. Θα πρέπει να δούμε το πρόβλημα από την άποψη τη Ένωση Κρατών που δεν έχουν αναγκαστικά τι ίδιε δυνατότητε, αλλά πρέπει να εργαστούν συλλογικά. Όταν εργαζόμαστε συλλογικά, μπορούμε αμέσω από την επόμενη μέρα να ε, διασφαλίσουμε την προστασία των πολιτών ή έστω ενό κράτου ή μια δυτική εταιρεία. Ευχαριστούμε κύριε Νέντ. Κύριε Τσεσνόφσκι, θέλετε το λόγο. Μπορεί το της εισηγητής να λέτε το λόγο. Όχι. Τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Πλασιβά. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Κάλφιν για την έκθεσή του αλλά και να τον συγχαρώ. Θέλω να τον ευχαριστήσω που έλαβε τον ευχαριστήσω που έλαβε υπόψη όλο το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι στιγμής, καθώς επίσης και τις ε, επικείμενες πρωτοβουλίες. Όλοι αναγνωρίζουμε ότι το διαδίκτυο παίζει σημαντικό ε, ρόλο στην οικονομία μας, στην κοινωνία μας, στην καθημερινή μας ζωή. Επίσης, οι κυβερνοαπειλές αυξάνονται και σε αριθμό και σε συχνότητα, αλλά και σε ε, περιπλοκότητα. Γι' αυτό είναι τα συστήματά μας όλο και πιο ευάλωτα. Χρειάζεται λοιπόν συντονισμένη προσέγγιση στρατηγική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ε, ανταποκριθούμε στις σημερινές προκλήσεις. Έχουν γίνει πολλά ήδη, αλλά απομένουν ακόμα περισσότερα για το μέλλον και θα ήθελα να επιβεβαιώσω την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταθέσει πρόταση ε, για μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια του διαδικτύου ε, το ε, τρίτο τρίμηνο του 2012. Έχουμε στόχο να φέρουμε μια συνολική και φιλόδοξη πρόταση. Ήδη εξετάζουμε ορισμένες από τις προτάσεις που ανέφερε ο κύριος Κάλφιν και ορισμένα αλλά αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέχρι στιγμής. Μεταξύ άλλων, η στρατηγική θα προβλέπει ένα ή περισσότερα νομικά μέσα και με τον τρόπο αυτό θα αποτελέσει σημαντικό βήμα αναβάθμισης από τη σημερινή ε, εθελούσια προσέγγιση σε μια πιο δεσμευτική. Παράδειγμα, νομικές διατάξεις που θα ορίζουν ε, συστήματα ανταπόκρισης σε έκτακτες ανάγκες σχετικά με τους υπολογιστές ή ε, κάποιες ε, υποχρεώσεις κοινοποίηση για τομείς εκτός των τηλεπικοινωνιών. Αναφέρθηκε ο τραπεζικός τομέας προηγουμένως, ίσως και ο ενεργειακός. Είναι όλες αυτές προτάσεις τις οποίες εξετάζουμε αυτό τον καιρό. Γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι για να επιτύχουμε στις προσπάθειές μας θα πρέπει να είμαστε συντονισμένοι σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή τα κράτη-μέλη να λαμβάνουν δράσεις και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους για τον ιδιωτικό τομέα, για την κοινωνία των πολιτών, αλλά και για το μεμονωμένο πολίτη. Τέλος, θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω τον κύριο Κάλφιν και όλους σας για την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση και να είστε βέβαιοι ότι θα ε, λάβουμε υπόψη στη στρατηγική μας ε, τις προτάσεις της έκθεσής σας. Ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το λόγο στον εισηγητή για να συνοψίσει. Παρακαλώ, αν να είστε σύντομος, γιατί έχουμε καθυστέρηση ήδη. Um. Ναι, θα είμαι σύντομο, Πρόεδρε, μην ανησυχείτε. Σα ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ του συναδέλφου, του Σκιώδη, τον κύριο Βανίστε Ρόι και του υπολείπου με του οποίου έχουμε συνεργαστεί για την έκθεση αυτή. Θέλω να ευχαριστήσω επίση πάρα πολύ του συναδέλφου για τα σχόλια που έκαναν τώρα. Κάποιε σύντομε απαντήσει στα σχόλια. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε αυτή τη συναντήληψη. το νέο επίπεδο της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο δεν θα αποτελέσει ένα άθροισμα των εθνικών συστημάτων, αλλά θα είναι ποιοτικό ε, άλμα για ένα πιο ασφαλές διαδίκτυο, το οποίο θα παρέχουμε ε, στους πολίτες και στις επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ε, ξεδιπλώνουν τις δραστηριότητές τους, να προσφέρουν τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στη στρατιωτική ασφάλεια και ε, την πολιτική ασφάλεια. Τι εννοώ. Περισσότερα κράτη-μέλη ε, μας είναι και κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ που αναπτύσσει τη στρατιωτική πτυχή ε, σε ένα κέντρο στην Εστονία για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Υπάρχει συνεργασία ήδη μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η στρατιωτική πτυχή. Εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο... Επικεντρωνόμαστε στην προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας, ε, πολιτικής φύσεως όμως, όχι στρατιωτικής και συνεργαζόμαστε και εμπρεόμαστε από τους μεγάλους μας εταίρους της ΗΠΑ. Πολιτείας. Βεβαίως έχουμε τις υπηρεσίες τραπεζικές, χρηματοπιστωτικές, υπηρεσίες υγείας. Όλα αυτά θα πρέπει να καλύπτονται από την ασφάλεια του διαδικτύου και χαίρομαι πάρα πολύ που και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε πρωτοβουλία ηγετική προς την κατεύθυνση αυτή και θα καταθέσει τη στρατηγική μετά τις ελληνές διακοπές για να έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε περισσότερο. Ε, περιμένω τις τροπολογίες των συναδέλφων. Η προθεσμία, δεν απατώμε, είναι η 5η Μαρτίου. Και θα χαρώ να συνεργαστώ μαζί σας για να ε, ολοκληρώσουμε την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Και μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι η 5η Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση Γκιουρκ. 20 μείζονες ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών και των επιχειρήσεων όσον αφορά τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Δίνω μέσα το λόγο στον εισηγητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να διαρθρώσω εδώ τα σχόλιά μου και να τα παρουσιάσω σε τρία τμήματα. Καταρχήν σχετικά με την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποτελεί τη βάση της σημερινής συζητήσεως και της γνωμοδότησης την οποία έχουμε καταρτήσει. Δεύτερον, θα ήθελα να αναφερθώ στη μεθοδολογία εργασίας την ε, οποία εφαρμόζουμε σαν Επιτροπή ε, και στην οποία συμμετέχουμε και τρίτον θα αναφερθώ λεπτομερώς στο περιεχόμενο του εγγράφου. Όσον αφορά το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, έφτασε νωρί σήμερα το πρωί, αλλά το θέμα της εκθέσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ένα από τα ε, σημαντικότερα θέματα ε, για το μέλλον που πραγματεύεται το Κοινοβούλιο, διότι προβλέπει ότι η πολίτες και η κοινή γνώμη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως διατυπώνουν την άποψη ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά που είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως τα τελευταία χρόνια. Το θέμα αυτό βέβαια δεν ε, μπορεί να διεκπαιρεωθεί ή να διατυπωθεί σε μία μόνο έκθεση. Δεν πρέπει ε, να ε, χαθούμε μέσα στη λεπτομέρεια και πρέπει να εξετάσουμε το σύνολο της εσωτερικής αγοράς, το οποίο όμως δεν έχει αντιμετωπιστεί με μία ενιαία μορφή μέχρι τώρα. Γι' αυτό και η Επιτροπή μας αποφάσισε να ασχοληθεί με ε, το γενικό πλαίσιο του θέματος. Έχουμε πολλές εκθέσεις, έχουμε ένα καλό σημείο εκκινήσεως. Η Επιτροπή βασίζεται εις τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρήσεων και του Volvit και από την άλλη πλευρά πρέπει να πούμε ότι από κοινού με τους συναδέλφους ευρωβουλευτές μπορούμε κατά πάσα στιγμή να ρουσιάσουμε πληροφορίες σχετικά με τέτοια θέματα και με τις αναλύσεις διότι τα θέματα αυτά απασχολούν τους πολίτες μας έχουμε μαζί τους διάφορες συζητήσεις και εδώ αναφερόμαστε εις την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να αντιμετωπίσει παραδείγματο παραδείγματος χάρη τις ε, προμήθειες υγειονομικού υλικού, το θέμα της ε, θέσεως σε κυκλοφορία των ε, αυτοκινήτων, την απονομή πτυχίων, τις αγορές μέσω του διαδικτύου. Υπάρχουν πάρα πολλές δυσχέρειες οι οποίες αναφέρονται στη την δυσλειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Και η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι η εξέλιξη είναι θετική διότι προσπαθούμε να διαρευνήσουμε αν υπάρχουν ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για το χώρο αυτό, εάν εφαρμόζονται Εάν ενδεχομένως μπορεί κανείς να πει ότι ο τρόπος λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει ε, νομοθετικό πλαίσιο ή ότι δεν υπάρχει σωστή εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου. Καταρτήσαμε λοιπόν έναν κατάλογο, δεν επαρκεί όμως αυτό, πρέπει να προτείνουμε και λύσεις για να ε, μπορέσουν να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα και γι' αυτό η ανάλυση αυτή αποτελεί ε, μία καλή βάση για να αναπτύξουμε την ε, έκθεση που έχουμε αναλάβει. Σχετικά με τη μεθοδολογία τώρα, θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθορίσει 20 θεματικές ενότητες και η Επιτροπή ΙΜΚΟ πρότεινε να επιλέξουμε ε, ένα τρόπο εργασίας όπου η αρμόδια επιτροπή θα αναλαμβάνει κάποια πτυχή. Ε, ε, έχουμε δηλαδή τρία θέματα για τα οποία εμείς είμαστε υπεύθυνοι. Το σημείο 14 είναι οι ε, ενεργειακές τιμές και οι λογαριασμοί. Μετά 16 όπου έχουμε ίδια αρμοδιότητα παράλληλα με την ε, Επιτροπή ε, ΙΜΚΟ και ε, υπάρχει επιπλέον η πρόσβαση σε χρηματοδοτικές δυνατότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η ΕΚΟΝ εμπλέκεται εδώ και στον τομέα αρμοδιοτήτων μας ε, περιλαμβάνεται η έκθεση αυτή διότι αναφερόμαστε στις κερατικές ενισχύσεις. Ε, σαν Κοινοβούλιο λοιπόν και Επιτροπή ε, μπορούμε να προχωρήσουμε αλλά πιστεύω ότι οι συστάσεις του Προέδρου της Επιτροπής ΙΜΚΟ μπορούν να αποτελέσουν την βάση ώστε ε, στη συνέχεια να μπορέσουμε και εμείς ε, να αναπτύξουμε τα θέματά μας και να προσεγγίσουμε τις απόψεις ε, των άλλων Ευρωβουλευτών και Επιτροπών. Εδώ λοιπόν ασχολούμαστε με τρία θέματα. Καταρχήν υπάρχει μία πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρέπει να δούμε ε, αν ε, είναι αποτελεσματική νομοθεσία, εάν έχει επιτύχει ή αν ε, ότι δεν έχει εφαρμοστεί επαρκώς η αν αυτό σε εθνικό επίπεδο. Το δεύτερο θέμα είναι η ε, θέμα λογιστικό και το θέμα των τιμών διότι οι τιμές έχουν φτάσει στα ύψη ε, στα προηγούμενα χρόνια ε, έχουμε δηλαδή μία αύξηση την οποία ατυχώς διαπιστώσαμε όλοι και ε, ε, πίσω από αυτή την αύξηση των τιμών κρύβεται η σημαντική αύξηση των τιμών των πρώτων υλών και λιγότερο η ε, απελευθέρωση του ανταγωνισμού. Δηλαδή ο ανταγωνισμός δεν ε, υπάρχει επαρκώ στην αγορά, αλλά βέβαια οι τιμές θα μπορούσαν να είναι ακόμη ψηλότερες. Δεν θέλω να σας πω δηλαδή ότι έχουμε προβλήματα σχετικά ε, με το θέμα αυτό. Υπάρχουν παράπονα των πελατών, τα βλέπουμε και στις εκθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι λογαριασμοί δεν είναι σαφείς ε, και υπάρχουν και πολλά άλλα προβλήματα τα οποία ε, δεν ε, βοηθούν στο να αντιμετωπιστεί το θέμα. Βέβαια δεν θέλω να σας πω ότι δεν χρειαζόμαστε ε, νέα νομοθεσία διότι το βασικό είναι ότι έχουμε 17 κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχουν εφαρμόσει το τρίτο πακέτο ενεργείας και αυτό είναι το πακέτο το οποίο θα διευκόλυνε πάρα πολύ το έργο και την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Γι' αυτό και θέλω να σας πω ότι πρόκειται για την εφαρμογή ε, της νομοθεσίας. Πρέπει να ενισχύσουμε και τις κυβερνητικές αρχές. Και τρίτον θέλω να αναφερθώ στα ε, έξυπνα δίκτυα, διότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε κανείς ε, να επωφεληθεί κανείς από τις δυνατότητες που μας δίνουν τα smart grids, τα έξυπνα δίκτυα αυτά και ε, ε, το σημείο 16 επίσης είναι της αρμοδιότητός μας διότι κυρία Πρόεδρε θα ήθελα να σας παρακαλέσω ίσως να παρακαλέσετε ε, να υπάρξει μεγαλύτερη ησυχία διότι εγώ δεν μπορώ να ακούσω τον εαυτό μου που μιλάω και δεν είναι δυνατόν κατά αυτόν τον τρόπο με τόσες, τόσο θόρυβο να μπορέσω να αναπτύξω την σκέψη μου. Σας παρακαλώ σταματήστε και λίγη ησυχία για να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα διότι διαφορετικά και για τον ομιλητή είναι δύσκολο να μπορέσει να σκεφτεί και να μιλήσει. Λοιπόν, επανέρχομαι λέει ο ομιλητής. Φτάνω στην κατάληξη, στο συμπέρασμα, δηλαδή στο σημείο 15 ποιότητα και μέση των ενεργειακών των ε, υπηρεσιών. Ε, εάν μπορούμε να ε, να μιλήσουμε για τις τιμές πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι διότι οι τιμές μειώνονται αλλά είναι απατηλή αυτή η μείωση των τιμών των ενεργειών της ενεργείας διότι ουσιαστικώς πρόκειται για διαρθρωτικά προβλήματα τα οποία έχουν ε, διαπιστωθεί. Υπάρχει μία διαδικασία παραβιάσεως που έχει ξεκινήσει κατά 15, 15 ε, κρατών που δεν έχουν εφαρμόσει τις διατάξεις ε, και όπου υπάρχουν παράπονα των πελατών και άλλων κρατών ε, για έλλειψη διαφανίας οι τιμές και τα τιμολόγια δεν είναι δυνατόν να συγκριθούν και πολλές φορές ε, ε, δεν προσφέρονται οι αντίστοιχες υπηρεσίες εις τους πελάτες και γι' αυτό οι πελάτες ε, παραπονούνται. Όσον αφορά τις διαρθρωτικές λύσεις, δηλαδή την εφαρμογή των νομικών διατάξεων και η δημιουργία ενός νέου θεσμικού πλαισίου, σκεφτείτε ότι, έχουμε να ψηφίσουμε και την έκθεση για την περιαγωγή, για το roaming, πέραν των προβλημάτων τα οποία πραγματεύομαι εγώ. Ε, πρέπει λοιπόν να υπάρξει μία επιτάχυνση της εφαρμογής των διαδικασιών. Θα χρειαστούμε ενδεχομένως και άλλα νομοθετικά μέτρα, αλλά πρέπει να ενισχύσουμε τις ε, κυβερνητικές ε, ε, διατάξεις και να υπάρξει μία διαφάνεια όσον αφορά τα έγγραφα. Επιπλέον ζητούμε πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντικές είναι κάτι το οποίο πρέπει να τονίσω ε, στην Επιτροπή μας και πρέπει να μπορέσουν να είναι σε θέση να σταθούν μέσα σε αυτή την κρίση και ως εκ τούτου πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διευκολύνουμε την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση μέσω δραστικών μέτρων. Δηλαδή είτε πρόκειται με την εφαρμογή κρατικών μέτρων ή μέσω ιδιωτικής χρηματοδότησης. Ε, ε, ε, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουν πρόσβαση στα, στην κοινωτική χρηματοδότηση και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ και στο γλωσσικό πρόβλημα και να προτείνω δύο λύσεις. Από τη μία πλευρά να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες και δεύτερον να δημιουργήσουμε ένα σύστημα one-stop shop, δηλαδή ε, ενιαίας αντιμετωπίσεως και ε, περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον τα σχόλια των συναδελφών. Των συναδέλφων. Ο κύριο Σενά. Λίγα λεπτά έχουμε για να αρχίσουμε τι ψηφοφορίε. Euh, Επιπλέον είναι δύσκολη στιγμή διότι κάποιοι μπαίνουν, κάποιοι βγαίνουν. Όμως ορισμένοι συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο. Ο κύριο Ενά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που σήκωσα τους τόνους, αλλά είναι πάρα πολύ δυσάρεστο και για τον εισηγητή, αλλά και για τους παρόντες από την αρχή της συνεδρίας. Συνεργαζόμαστε σε τέτοιες συνθήκες. Δεν ακούγαμε τίποτα γιατί θέλουμε να ακούμε τη διερμηνία σωστά και να μπορούμε να κάνουμε σχόλια, επειδή δεν έχουμε χρόνο. Δύο βασικές ανησυχίες για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις. Ποιες είναι για τους πολίτες, πρώτον. Κοιτάξτε, Εγώ δεν έχω πρόσβαση στα κέντρα δημοσκόπησης, αλλά ο κόσμος στο δρόμο μιλάει για την απασχόληση και για την αγοραστική δύναμη. Μα αυτό μας αφορά άμεσα. Και οι επιχειρήσεις είναι θύμα του αθέμητου ανταγωνισμού, μείωση της δραστηριότητάς του και δυσκολίες. Και ε, αργοπεθαίνουν γιατί ε, δεν ε, έχουν και πρόσβαση στη δανειοδότηση. Βλέπουμε τις τρεις κατηγορίες. Υπηρεσίες ίντερνετ, τηλεφωνία, ενέργεια, χρηματοδότηση μπορούμε να συνοψίσουμε. Στο πρώτο, στην ενέργεια, και ερδοσκοπία όσο παρα... καταναλώνουμε περισσότερη ενέργεια από ό,τι παράγουμε, θα έχουμε πρόβλημα γιατί γίνεται κερδοσκοπία. Ορισμένοι εσχροκερδούν και πλουτίζουν χωρίς να παράγουν. Ε, υπηρεσίες διαδικτύου, τηλεφωνία στη Γαλλία ήρθε ένας νέος φορέας και έδειξε ότι υπήρχε αθέμητη συμφωνία μεταξύ των μεγάλων ομίλων που έχουν αστρονομικά κέρδη στην πλάτη των καταναλωτών. Και τέλος, για τη χρηματοδότηση και την οικονομική στήριξη θα ήθελα να επιμείνω στον ειδικό ρόλο των τραπεζών. Οι τράπεζες που τις διέσωσαν τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση και αρνούνται σήμερα συστηματικά να βοηθούν ε, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν είναι σπάνιο να βλέπει κανείς ανθρώπους που έχουν επενδύσει τα πάντα στην εταιρεία τους να χάνουν μέσα σε λίγες εβδομάδες τον καρπό ενός ολόκληρου ε, βίου ε, εργασιακού γιατί τους αρνούνται ένα πολύ μικρό δάνειο οι τράπεζες. Ευχαριστώ κύριο Ζρουμπίχη. Äh, Ζητώ συγγνώμη, λέει κύριε ε, Ρεμπίχ, για την καθυστέρηση. Θέλω να συγχαρώ τον συνάδελφο Γιώργ. Ακούμε πραγματικά τι απασχολεί τον κόσμο και είναι απόλυτη προτεραιότητα αυτό το θέμα. Η κρίση χρέους καταλήγει σε μια συζήτηση πώς κάνουμε μεταφορές πιστώσεων από τον Α στο Β. Αυτό σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ επιπόλαια η προσέγγιση μας. Δεν μπαίνουμε στο βάθος ε, της υπόθεσης. Έχουμε χιλιάδες νέους ανέργους στο δρόμο και θα πρέπει να δούμε πώς θα κάνουμε τους νέους μας άνδρες και γυναίκες να ιδρύουν επιχειρήσεις για να καταπολεμηθεί η ανεργία. Γι' αυτό καλό και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δραστηριοποιηθεί περισσότερο εδώ. Χρειαζόμαστε κίνητρα οι νέοι μας και οι νέες μας να επιδείξουν επιχειρηματικό πνεύμα και να δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις απασχόλησης. Αυτό σημαίνει θα πρέπει να έχει και καλά κέρδη η επιχείρηση και να είναι εποφελής και για τις δύο πλευρές. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γιώργ που ε, ασχολήθηκε με αυτό το τόσο σημαντικό θέμα και μας έκανε τόσο καλές προτάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Δεν έχω κανέναν πλέον εγγεγραμμένο στη λίστα, στον κατάλογο με του ομιλητέ, Ο λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εάν υπάρχει κάποιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κανεί δεν βρίσκεται εδώ. Εάν ο εισηγητή θέλει να προσθέσει κάτι... Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τους συναδέλφους για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους και πάλι να σας επιστήσω την προσοχή ότι είμαστε σε επαφή με την καθήλια αρμόδια επιτροπή που είναι ε, της εσωτερικής αγοράς ε, και των καταναλωτών, ΙΜΚΟ, και είπαμε ότι σε αυτά τα τρία θέματα είμαστε εμεί αρμόδιοι και έχουμε στη δική μας γνωμοδότηση ε, άποψη. Για αυτά τα θέματα μπορείτε να κάνετε τις απολογίες σας μέχρι τις 12 Μαρτίου. Στη συνέχεια θα επεξεργαστώ τις απολογίες και θα τις βάλω και στο κείμενο της έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, ε, Ευχαριστούμε κύριε Γιούρκ. Θυμίζω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών λίγη στις 22 Μαρτίου 2012 το μεσημέρι. Ετοιμαστείτε λοιπόν για τις ψηφοφορίες που θα ξεκινήσει σε δύο λεπτά.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 Εάν θέλετε, καθίστε για να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες. Το λόγο, όμως, έχει ζητήσει ο κύριος Ρόντ. Του δίνω το λόγο και αμέσως θα περάσουμε στην ψηφοφορία. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο θέματα ήθελα να θέσω. Φτάνοντας σήμερα το πρωί, είδα διαφημιστικά πανό εδώ απ' έξω. Ολόκληρη διαδήλωση μπροστά από την αίθουσα. Ορισμένοι προβάλλονται ως ήρωες της πράσινης ενέργειας και άλλοι πάλι πολέμοι της οικολογικής παραγωγή ενέργειας. Σκοπεύω να απευθύνω επιστολή στον Πρόεδρο, έτσι ώστε στο μέλλον να μην έχουμε τέτοιες διαδηλώσεις ε, ε, έξω από την αίθουσα. Τι είναι αυτές οι αφήσει, τι είναι αυτές οι εκδηλώσεις. Εμείς ερχόμαστε το πρωί εδώ να εργαστούμε. Αυτό ήταν το πρώτο. Έρχομαι τώρα στην ψηφοφορία. Βλέπετε τον κατάλογο ψηφοφορίας σε δύο από τις εκθέσεις θα ψηφίσουμε για να δούμε εάν θα δώσουμε ή όχι διαπραγματευτική εντολή στον εισηγητή μας. Ενώ για τους άλλους δεν υπάρχει διαδυνατότητα. Μπορεί αυτό να συμφωνεί με τον κανονισμό ή με τους κανόνες που ισχύουν στην Επιτροπή μας. Αν θέλουμε μπορούμε να ψηφίσουμε για να δώσουμε ή όχι διαπραγματευτική εντολή, στον εισηγητή, αλλά νομίζω ότι είναι καινοφανής αυτή η πρακτική και η διαδικασία. Τα τελευταία δυόμιση χρόνια, κάθε φορά που ψηφίζαμε, εγκρίναμε την έκθεση δηλαδή, αυτό θεωρείται αυτόματα ε, ως διαπραγματευτική εντολή προς τον εισηγητή. Αν θέλουμε τώρα να αλλάξουμε τη διαδικασία, θα πρότεινα να πούμε ότι θα πρέπει κάθε φορά να ψηφίζουμε για τη διαπραγματευτική εντολή. Και όχι επιλεκτικά για ορισμένες εκθέσεις, αλλά για όλες. Αλλιώς κινδυνεύουμε ε, η ψηφοφορία αυτή να καταλήξει σε νέες πολιτικές μάχες. Δηλαδή δεν θα έχουμε μόνο την παράθεση επί της ουσίας πολιτική, αλλά θα κάνουμε και συνδικαλισμό. Ε, ποιος είναι ο εισηγητής, μήπως είναι πράσινος, α, χρειάζεται διαπραγματευτική εντολή να την ψηφίσουμε χωριστά, αφού ψηφίσαμε την ουσία της έκθεσης. Αυτά τα πράγματα δεν είναι ε, αντάξια μια σωστή κοινοβουλευτική λειτουργία ούτε αξιοπρεπή. Για να γνωρίσουμε λοιπόν εάν θέλουμε να δώσουμε διαπραγματευτική εντολή στον εισηγητή μας, θα πρέπει να ξέρουμε με ποιο τρόπο θα το κάνουμε να αφορά όλες τις εκθέσεις και όχι μόνο ορισμένες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πριν δώσω το λόγο σε όσου τον ζήτησα, να δώσω δύο απαντήσει στον κύριο Ροντ. Πρώτον, ότι καλέσαμε την Υπηρεσία Ασφαλεία και ήδη αυτό που έγινε έξω από την αίθουσα διαλύθηκε. Και Έπειτα και οι τρεις εκθέσεις θα ψηφιστούν. Και θα κάνουμε αυτό που κάναμε πάντοτε. Ο κύριος Μπουτικόφερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα μόνο να πω κάτι για αυτή τη μικρή δράση έξω από την αίθουσα. Σε καμία περίπτωση με ενόχλησε μένα αυτό. Εγώ μπορεί να μην δοξάστηκα ως ήρωας, Πράγμα που μπορεί κανείς να θεωρεί λυπηρό, αλλά ε, με ενθάρρυναν να διαπιστώσω και να ε, καταλάβω ότι μπορεί κάποιος να γίνει ήρωας και εντός του Κοινοβουλίου. Και παρακαλώ αυτό μην το θεωρείτε ενόχληση, απλώς ως ε, φιλική ενθάρρυνση. Και με αυτή την περιορισμένη έννοια θα ήθελα αγαπητέ συνάδελφοι να διαφωνήσω μαζί σας. Ευχαριστούμε κύριο Ρόιλ. Κύριε Μπιουτικόφερ, αγαπητέ συνάδελφε, θέλω να διαφωνήσω κατηγορηματικά μαζί σας. Έχει δίκιο ο κύριος Ρόντε. Γιατί όταν έξω από το κοινοβούλιο, ακόμα και μέσα στο κοινοβούλιο και έξω από μια αίθουσα που ψηφίζουμε, λαμβάνει χώρα μια πολιτική δράση, ανεξάρτητα από τη δράση, που ε, παίρνει θέση και προσπαθεί να επηρεάσει τα πράγματα, αυτά τα θέματα δεν έχουν καμιά θέση στο Κοινοβούλιο. Εσεί συνήθω είστε τόσο επικριτικό στα λόμπι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείτε. Θεωρώ ότι είναι ανεπίτρεπτο κάτι τέτοιο και ευχαριστώ πάρα πολύ που έχετε λάβει δράση. Αλλιώ, σε λίγο μπορούμε να έχουμε και μεγάλες εταιρείε ενέργειας που να κρεμάνε πανώ έξω από την πόρτα μας. Παρατήρηση δεύτερη, διαδικαστική αυτή κύριος Κόφερ εκτό μικροφώνου δυστυχώ δεν ακούγεται. Κοιτάξτε, το κοινοβούλιο είναι ένας χώρος που ε, παραμένει ελεύθερος ε, τέτοιων ε, δραστηριοτήτων. Αλλιώ μπορούμε κάθε μέρα να διοργανώνουμε και πανηγύρια εδώ πέρα μέσα. Είναι κακό αυτό το παράδειγμα και το προηγούμενο. Δεύτερη παρατήρηση. Σωστά είπε ο κύριος Ρότε ότι συνήθως η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Κυρίες και κύριοι, σα ενοχλώ πάρα πολύ στις ιδιωτικέ συνομιλίε. Πείτε το μου να σταματήσω. Λοιπόν, η συνήθι κανονική διαδικασία είναι να αποφασίζει η Επιτροπή και πάει σε πρώτη ανάγνωση μετά αυτό στο Κοινοβούλιο, στην Ολομέλεια, έτσι ώστε όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου να έχουν την ευκαιρία να ψηφίσουν και να πούν τη γνώμη του. Και από εκεί και πέρα γίνεται διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο. Αυτή είναι η κανονική διαδικασία. Ακριβώς όμως επειδή είναι κανονική διαδικασία, είπε ο κύριος Ρόντε, στην περίπτωση που χρειάζεται διαπραγματευτική εντολή ε, προς τον εισηγητή να διαπραγματευτεί εκ των προτέρων, ε, γίνεται αυτό στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή και έχει δίκιο να μην είναι έκτακτη αυτή η δραστηριότητα και η διαδικασία να είναι πάγια. Εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός ε, και επικριτικός απέναντι στις συμφωνίες πριν την πρώτη ανάγνωση. Ε, δίνει τη δυνατότητα αυτό σε ένα, δύο ή τρεις συναδέλφους, ανεξάρτητα από το ε, αν είναι καλή, κακή, σωστή ή λάθος, η πρόεδρο διακόπτει τον ομιλητή. Λοιπόν, δίνει την ευκαιρία μόνο σε δύο-τρει ε, βουλευτέ να επηρεάσουν τα πράγματα και οι υπόλοιποι που δεν είναι μέλη τη Επιτροπή μα έχουν μηδενική ευκαιρία. Διότι απλώ του ε, ανακοινώνεται ένα αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο που μπορούν να πούν ναι ή όχι σε αυτό. Άρα θα πρέπει να γίνεται μια διάκριση ανάμεσα στα πολιτικά σημαντικά ζητήματα που πρέπει να αποφασίζει η Ολομέλεια ή διαδικασίες που είναι απλώς συνέχιση ε, παρελθούσης ε, δραστηριότητας. Ας πούμε, για το roaming, την περιαγωγή, ε, μας πιέζει ο χρόνος, υπάρχει προϊστορία και απλώς συνεχίζεται. Θα πρέπει να συνεννοηθούμε αν το θέλουμε δεν το θέλουμε, για το roaming επαναλαμβάνω είναι μεγάλη χρονική πίεση, η πολιτική απόφαση επί της αρχής έχει ήδη ληφθεί, αλλά για το άλλο είναι τελείως λάθος. Οι συνάδελφοι που δεν είναι μέλη της Επιτροπής μας δεν έχουν ε, την ευκαιρία να εκφραστούν και αυτό δεν είναι δημοκρατικό. Ευχαριστούμε κύριε Ρόιλ. Ο κύριος Τούρμες έχει ζητήσει το λόγο και μετά από αυτό θα έλεγα ίσως να ξεκινήσουμε την ψηφορία. Κύριε Τούρμες. Uh, uh, Όταν έχουμε σημαντικές ψηφοφορίες, είναι μεγαλύτερη συναισθηματική φόρτιση ε, εντός της αιθούσης. Και έχουμε σημαντική ψηφοφορία και για την ενεργειακή αποδοτικότητα και για την περιαγωγή και για τη διαφάνεια ε, στις συμβάσεις ε, έκθεση Καρίνς. Η συζήτηση τώρα είναι για την εντολή ή όχι. Χτες μία ώρα το συζητούσαμε στους συντονιστές αυτό το θέμα. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να επανέλθουμε κάποια στιγμή σε αυτό, αλλά προς το παρόν... Προς το παρόν... Και για να εξασφαλίσουμε ε, ομαλή και κανονική ψηφοφορία ως εισηγητής για την ε, ενεργειακή αποδοτικότητα θα παρακαλούσα να ψηφίσουμε για την περιαγωγή και σιγά σιγά με τη σειρά να πάμε στην επόμενη οδηγία και να ψηφίσουμε και αυτή. Χρόνο δεν έχουμε τώρα να κάνουμε συζήτηση επί της αρχής για το αν θα δοθεί διαπραγματευτική εντολή ή όχι. Ευχαριστώ πολύ. Σας λέω πάντως ότι καταρχήν συμφωνώ με τη θέση του κυρίου Ρόντε, αλλά ε, προς όφελος της σωστής, ε, της καλής ψηφοφορίας, παρακαλώ να περάσουμε μέσα στη ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Ε, Θα ήθελα να ξεκινήσει η ψηφοφορία. Ο συνάδελφος Ούντλερ θέλει το λόγο. Ή συνάδελφος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να σέβεται κανείς και τον εαυτό του, πάνω απ' όλα δεν είναι δυνατόν στις 10 να μας δίνονται τα έγγραφα για μια τόσο σημαντική ψηφοφορία Την προηγούμενη, το προηγούμενο βράδυ στις 10. Θα πρέπει κανείς να έχει αρκετό χρόνο στη διάθεσή του για να μπορεί να μελετάει και τα έγγραφα για την ψηφοφορία. Κυρία Πρόεδρε, προσέξτε παρακαλώ περισσότερο το θέμα αυτό, να υπάρχει χρόνος μεταξύ της ε, διανομής των ε, εγγράφων και τη ψηφοφορία. Δεν μπορεί κανεί να ξενυχτάει για να διαβάσει τα έγγραφα που του δόθηκαν μόλι το προηγούμενο βράδυ. Πρόεδρο, έχετε δίκιο, μάλιστα. Το σημειώνουμε. Ξεκινάμε με την περιαγωγή. Η κυρία Νίμπλερ έχει δει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης ηγητές. Εβδομάδες ολόκληρες ψάχναμε συμβιβασμούς που να μπορούν να γίνουν δεκτοί από μεγάλη πλειοψηφία του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά όλους τους συναδέλφους που εργάστηκαν πάρα πολύ επικοδομητικά. Δεν υποστηρίζονται όλοι οι συμβιβασμοί μένα από όλες τις πολιτικές ομάδες, αλλά πρέπει να σας πω ότι ήταν υποδειγματική η συνεργασία και ευχαριστώ και πάλι τους συναδέλφους. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Άρθρο 1. 115 και 116 τροπολογίες μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 117. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 30. Ήμκο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 121. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. από κοινού 122, 32, 11. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 127. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Από κοινού 128, D. Με συγχωρείτε, προηγουμένω ΣΥΜΚΟ 34. Υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Από κοινό κατάλογο των τροπολογιών από το 12D ως το 35D. Υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Από κοινό 134-135. Υπέρ, κατά, αποχέ. εγκρίνεται. 137 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές μοιάζει να απορρίπτεται. Αλλά ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για να είμαστε βέβαιοι. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Πάλι, ό,τι και να κάνουμε, ένας από το είναι επιπλέον. Τώρα είναι εντάξει. Πέρα τη προφοριες εγκρινεται Εγκρίνεται. 32-26. 116. Όχι, 16 υπέρ. Με συγχωρείτε. Σφάλμα. Κομπρομίσο 3. Αφαβόρε. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος μάλλον. Έλεγχος για το 17. Αλλά το τούτη... Δεν να απαντές. Πέρας της ψηφοφορίας. Πέρας. Και πάλι είναι παραπάνω δύο από το ΕΛΚ. Ένας. Κάποιος περισσεύει πάντως. Ένας από το ΕΛΚ είναι παρα, παραπάνω. 30-26. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε. Ας ελέγξουμε. Πέντε. Εψήφισαν απαντές. Πέρας. Απορρίπτεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 202 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Από κοινού 224, 225 και 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 226 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 240. 241 και 50 από κοινό υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 243-244 από κοινού υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Οι 100 και η 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 245 υπέρ. Με συγχωρείτε, 34 προηγουμένως. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 245 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10. Συμβαστική πρόταση 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 251 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 263 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 265 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 56 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 280 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 281 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 282 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 283 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 296 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 299 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 303 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 304 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 41 και 305 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 324. υπέρ.

325 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 326 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 50, 338 και 72 από κοινού. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 72. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ήμκο. 74. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 341. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 343 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβεβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 359 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ήμκο 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 73 υπέρ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 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Από κοινού 1 και 10 και 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 80 τροπολογία 80 Και την 78, μάλιστα. 78, υπέρ. Κατά τη δική μου τη γνώμη 80 ήταν. Λοιπόν, 80 υπέρ. Κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 82 υπέρ. Κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ήμκο 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 89 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. Super. Άρχεται η ψηφοφορία. Πάλι είναι δύο υπεράριθμα τα μέλη του ΕΛΚ. Io il mio l'ho tolto perché... Ancora ούνα. Ένα είναι πάλι παραπάνω. Okay. 35... 35 προς 20. Εγκρίνεται. 91. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 94. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 99 και 100 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6, 20, 108, 109 μαζί. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 111 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 112 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 114 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 24 ε, συγγνώμη υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ονομαστική. Aperta la Άρχεται η ψηφοφορία. Πάλι είναι δύο τα μέλη του ΕΛ που είναι Φύγαν. Όλα εντάξει. Πάλι όχι. Πάλι είναι δύο υπεράριθμα τα μέλη του ΕΛΚ. Δύο τα μέλη του ΕΛΚ που περισσεύουν φύγαν ή όχι. Ένας έχει μείνει. Ωραία. Έχουμε αποτέλεσμα. 54 υπέρ, 5 κατά εγκρίθηκε. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία. Συγχαρητήρια στη συνάδελφο Νίμπλερ. Περνάμε εάν συμφωνείτε, να συνεχίσουμε, να ξεκινήσουμε μάλλον τι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο. Αυτό είναι το αντικείμενο τη ψηφοφορία. Κατά πόσον θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο. Ηλεκτρονική ψηφοφορία υπέρ. Μάλλον άρχεται η ψηφοφορία. Πάλι είναι δύο τα μέλη του ΕΛΚ που περισσεύουν. Κάποιοι αναπληρωτέ σα βγάλουν την κάρτα του. Πάλι μένει ένα. Ναι. Εντάξει τώρα, ωραία. Αποτέλεσμα. 46 υπέρ της έναρξης διαπραγματεύσεων, άμεσων διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Ευχαριστούμε. 46 προς ένα. Ευχαριστούμε τη συνάδελφο Νίμπλερ. Κύριε Τούρμες, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μετά από έξι μήνες ε, εντατικής εργασίας σήμερα θα ψηφίσουμε ε, την ε, έκθεση για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω όλες τις επιτροπές ε, για την καλή συνεργασία και θέλω να σας πω στο προσωπικό μας ότι ερισμένοι εξ αυτών όχι μόνο την εβδομάδα αλλά και τα Σαββατοκύριακα πέρασαν να προετοιμάζουν τους ε, καταλόγους ψηφοφορίας για τις τροπολογίες. Αφού συζήτησα με την Πιλάρ και άλλους συναδέλφους του ΕΛΚ αποφάσισα να αποσύρω την τροπολογία 59 η οποία ήταν μία τροπολογία που δημιουργούσε προβλήματα στο ΕΛΚ για την τελική ψηφοφορία, οπότε το δέχομαι και αποσύρω αυτή την τροπολογία. και κατόπιν αυτού μπορούμε να ξεκινήσουμε κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Τούρνς, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε μία πολύ μακρά ψηφοφορία και γι' αυτό ελπίζω να υπάρξει καλή συνεργασία. Καταρχήν τροπολογία 120. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται τροπολογία παρακαλώ αυτούς τους οποίους δεν θέλουν να ψηφίσουν να εγκαταλείψουν την αίθουσα όπως και οι συνεργάτες οι οποίοι θορυβούν πολύ. Τροπολογία 331 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 333 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Έλεγχος για την 333 ηλεκτρονικός ε, ξεκινά. Έχουμε δύο ΕΛΚ επιπλέον και παρακαλώ ακόμη έναν συνάδελφο να τραβήξει την κάρτα του. Τώρα είμαστε εντάξει. Ψήφισαν η κυρία Μαντουρέλ. Κύριε Πρόεδρε τι θα γίνει με το ΕΛΚ. Ε, ε, ψηφίζουν δύο παραπάνω. Ε, όταν ψηφίζουμε με το μηχάνημα είναι εντάξει, αλλά όταν ψηφίζουμε με ανάταση της χειρός ε, μπορεί να μην τους βλέπετε. Δεν μπορούμε να το λύσουμε αυτό το θέμα διαπαντός τώρα. Ευχαριστώ. Κύριε ε, δεν μπορούν δύο υπεράριθμοι να επηρεάσουν τόσο πολύ την όραση κάποιου και να τον κάνουν να μην διακρίνει. Συστηματικά περσέβουν δύο. Παρακαλώ βγάλτε τις κάρτες σας, αλλά παραμείνετε στην αίθουσα, γιατί μπορεί κάποιος να χρειαστεί να φύγει. Λοιπόν, δύο αναπληρωματικά μέλη που παρίσταται παρακαλώ να μην ψηφίζουν συστηματικά, αλλά να μην φύγουν κιόλας γιατί μπορεί να χρειαστεί να ψηφίσουν. Καλά, ε, ε, αν είναι δύο παραπάνω δεν σημαίνει ότι η πρόεδρος δεν τους βλέπει και χάνει την όρασή της. Passiamo allora per quanto riguarda, grazie, l'emendamento 3 για την ε, τροπολογία 333 η οποία περίφθη προχωράμε στην 337, 38 και 39 μαζί ε, ταυτόσιμες τροπολογίες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται τροπολογία 341 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Θέλετε να ελέγξουμε. Όχι. Για το δεύτερο τμήμα τότε. Δεν υπάρχει. 343 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 344 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 346 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται ηλεκτρονικός έλεγχος λίγη 28 επί, υπέρ 29 κατά περίφθη αλλά ίσα ίσα η κυρία Φόρντ Με συγχωρείτε, δεν πίεσα γέρο στο το κουμπί μου, οπότε θα είχα υπερψηφίσει. Μπορούμε να ξαναελέγξουμε. Ναι, αλλά είμαστε 29-29, οπότε και πάλι θα είχε απορριφθεί. Λοιπόν, απερίφθη 346 λαμβάνοντας υπόψη ε, την ψήφο της κυρίας Φόρ που υπερψήφισε αλλά και πάλι θα ήμασταν 29 προς 29 349 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται σε μαζί οι 350-352 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ηλεκτρονικός έλεγχος Ξεκινά. Λίγη. Τριάντα ένα υπέρ, 27 κατά. 357 εγκρίθηκε. Με συγχωρείτε, 352 λέει πρόεδρος εγκρίθηκε. Περνάμε στην 357. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν σηκώσατε καλά τα χέρια σας. Ε, ηλεκτρονικός έλεγχος. Για την 357. Εγώ νομίζω ότι υπερψηφίστηκε, αλλά για να δούμε. Λίγη ψηφοφορία. 41 υπέρ, 17 κατά. Αλλά δεν είχαν σηκώσει 41 τα χέρια τους πριν. 358 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Και πάλι ηλεκτρονικός έλεγχος για 358. Ξεκινά. Λίγη. 26 υπέρ, 32 κατά, απερίφθη η 358. 365 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 363 362 με συγχωρείτε λέει η πρόεδρος υπέρ 362 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι ενεκρίθη, αλλά πάλι δεν βγάζουμε άκρη με τα χέρια. 362 ηλεκτρονικός έλεγχος. Λίγοι. 43 υπέρ, 16 κατά. 368 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται 9 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται 375 υπέρ κατά Αποχέ απορρίπτεται 374 υπέρ κατά απόχέ απορρίπτεται 373 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 373. 373 ηλεκτρονικός έλεγχος. Έληξε. 26 υπέρ, 32 κατά, απερίφθη. Η 372. 372 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 380 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ηλεκτρονικός έλεγχος για 380. 28 υπέρ 30 κατά απορρίπτεται 378 υπέρ κατά σχετικά με την σχετικά με 377 ηλεκτρονικός έλεγχος. 378 είναι, ε, με συγχωρείτε, αλλά υπάρξει κάποια σύγχυση. Για την 378, την τροπολογία 378 ξεκινά ηλεκτρονικός έλεγχος. έχουμε έναν φιλελεύθερο πλεονάζοντα αυτή τη φορά. Λοιπόν, 378, 43 υπέρ, 16 κατά, ε, άρα ενεκρίθη. 377 τώρα, υπέρ. Σηκώστε τα χέρια όσοι είστε υπέρ, κατά αποχές απερίφθη. Ηλεκτρονικός ε, έλεγχος 377 ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη. 31 υπέρ 29 κατά ενεκρίθη. Είναι τόσο μικρές οι διαφορές ώστε είναι πολύ δύσκολο να το ξεχωρίσει κανείς. 379 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, ας ελέγξουμε και πάλι εγώ νομίζω ότι ενεκρίθη και χρειαζόμαστε να ψηφίσουμε 376 υπάρχει ένα σχόλιο Λοιπόν, το 377 ε, ψηφίστηκε και η γραμματεία λέει και λέγει ότι το 77 και το 76 καταπίπτουν. Και αυτή είναι η απάντηση προς τον κύριο Ρούμπικ σχετικά με το 379 λίγη ηλεκτρονική ψηφοφορία. 28 υπέρ, 29 κατά. Απερίφθη. Καταλαβαίνετε με τέτοιες μικρές διαφορές γιατί είναι δύσκολο να μπορέσει κανείς να το κρίνει από την ανάταση χειρών. Περνάμε τώρα στο 381. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 382-383 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά ένβη 26 υπέρ κάναμε το 6 την 6 και τώρα είμαστε στην 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 399 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 402 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 404 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 403 και 406 μαζί, υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος, ξεκινάει η ψηφοφορία για την 403 και 406 μαζί. Λίγη ε, ενεκρίθη 41 ε, ψήφους υπέρ. 409 ε, μέχρι την 27 εγκρίνεται 413 υπέρ κατά είμαστε στην 413 επαναλαμβάνω υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 414 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 412 Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 414. Λίγη ηλεκτρονική ψηφοφορία 33 υπέρ 25 κατά Εγκρίνεται Η 414 <clears throat> Ενεκρίθη Και περνάμε τώρα στην 412 Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 416 και 417 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 418 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 419 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 420 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 423 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 423 ξεκινά Λίγοι. 27 υπέρ, άρα απορρίπτεται. Η 423 συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 116 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 1473 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1475 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1477 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ηλεκτρονικός έλεγχος στη 1477. Λίγοι. 29 a favore, 30 contrario. Απερίφθη. 774 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη. Απερίφθη. Με 22 υπέρ 35 κατά. 628 υπέρ κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά α, αποχές απορρίπτεται. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Η συμβιβαστική 3 υπερψηφίστηκε αλλά κοιτάμε σε ποια σελίδα πρέπει να μετακινηθούμε και πάμε τώρα στη συμβιβαστική 4. Ε, η 3, ε, τι έγινε, εγκρίθηκε λέει η πρόεδρος η συμβιβαστική τροπολογία 3. Ενεκρίθη, ενεκρίθη, δεν χρειάζεται να την ελέγξουμε. Θα ήθελα να δω ποια είναι η έκβαση αυτής της ψηφοφορίας. Λοιπόν, ε, θέλετε να ξέρετε ποιος ψήφισε τι. Ξεκινά ψηφοφορία για τη συμβαστική τρία. για να ικανοποιήσουμε την περιέργεια. Λίγοι. 48 υπέρ, 8 κατά. Ενεκρίθη. Τώρα πάμε στη συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά. 115 μετά από τη συμβιβαστική 4 είμαστε στην τροπολογία 115. Την ε, εντοπίσατε υπέρ, κατά. Αποχές ενεκρίθη. 117 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά. Αποχές ενεκρίθη. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος σχετικά με το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 117. Ξεκινά. Λίγη. 26 υπέρ, 33 κατά, απερίφθη. Αυτή τη φορά είχατε δίκιο. Συμβιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η ε, τροπολογία 39 του περιβάλλοντος. NV39 στη σελίδα 25. 24 προς 25 μάλλον την ε, βρήκατε. MV39 και θα ψηφίσουμε μόνο το δεύτερο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές ενεκρίθη. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ξεκινά. Λίγη. 42 υπέρ 17 κατά ε, ενεκρίθη. Συμβιβαστική 6 είναι περίπου στη σελίδα 28-29. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Για τη συμβιβαστική 6 σελίδα 29. Λίγη. Απερίφθη. Ε, 27 υπέρ, 32 κατά. Εγώ έκανα λάθος. Ε, η 6α, συμβιβαστική 6α υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7. Σελίδα περίπου 33. 33 κάτω. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε περίπου στη σελίδα 40 στην τροπολογία 23. Την βρήκατε Ε, τροπολογία 29 και 110 μαζί. Έχετε βρει που βρισκόμαστε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Λίγη ψηφοφορία. Απερίφθη. Τροπολογία 739 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι ενεκρίθη, αλλά ελάχιστοι σήκωσαν τα χέρια του. 739, τροπολογία 739. Ξεκινά. Νομίζω ότι εγκρίθηκε. Λίγη. 35-16 ενεκρίθη. Υπάρχει και μια προφορική τροπολογία. Η 705 με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 698 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 707 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 789 ε, στη σελίδα 47 <clears throat> υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος ξεκινά. Ένας πλεονάζων, ένα ΕΛΚ πλεονάζων, με συγχωρείτε. Ακόμη ένας βουλευτής του ΕΛΚ πλεονάζει. Λίγοι. 27 υπέρ, 32 κατά, απερίφθη. Συμβιβαστική 8 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Σελίδα περίπου 56 391 και 25 σελίδα 56 ε, υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος Λίγη. Ενεκρίθη. 51 υπέρ και 7 κατά. 392 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 393 υπέρ. Για 392 θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο. το Λίγη ψηφοφορία, 27 υπέρ, 32 κατά, περίφθη. 393 τροπολογία υπέρ. Κατά. Απερίφθη. Συμβιβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές ενεκρίθη. Τώρα περνάμε στη συμβιβαστική 10, περίπου σελίδα 70. Συμβιβαστική 10. Ε, βρήκατε τη συμβιβαστική 10 στην ε, σελίδα 70. 67-70. Perfetto. Compromesso 10 a favore. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα περνάμε περίπου στη σελίδα 88. 87-88. 1677 και 1679. Βρήκατε ε, πού ακριβώς είναι αυτές οι, αυτές οι τροπολογίες. 84-88 σελίδα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Απερίφθη αλλά να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο ε, σχετικά με την 1777-79. Ε, Λίγη ψηφοφορία. 27 υπέρ, 31 κατά, απερίφθη. 1778 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Και τώρα, σε μπλοκ, 1321, 22, 23, 24, 1400, 80-81 on block από κοινού. Νομίζω ότι on block. On block. 90. Λίγο πολύ στη σελίδα 90. Βλέπω εγώ, σε άλλους 87. 1321, 1322, 1323, 1324, 1781, 1780. Το βρήκατε όλοι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1782, 1783. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος. 1782-83. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 29 προς 30. Απορρίπτεται. Είχατε δίκιο που θέλατε να ελέγξουμε. 1325 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 1326 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 1328 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1327 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος για το 1327 άρχεται η ψηφορία. πέρας 32 προς 26. Εγκρίνεται. 1329. Άρχεται η ψηφοφορία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 59 έχει αποσυρθεί. 60. Υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος πέρας 29 προς 30 απορρίπτεται Compromesso 12. Συμβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 13. Σελίδα 93 ή 95. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. «826 Τόμσεν, υπέρ» κατά, αποχές, εγκρίνεται. 775 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17. Έλεγχος. Για την 777. 75, συγγνώμη. 775. Έλεγχος. πέρας 24 προς 33 απορρίπτεται 14 τροπολογία 14 υπέρ κατά έλεγχος Votazione chiusa. 25... 25 προς 32. Απορρίπτεται. Emendamento 17 a favore. Contrari. Approvato. Compromesso 14. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 15. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. 1472 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. 1472. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 29 προς 30. Απορρίπτεται. Απορρίφθηκε 1472. 78 και 91 μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 28 προς 29. Απορρίπτεται. ...92 και 118 από κοινού. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Έλεγχος. 92-118 από κοινού. 34 προ 25 εγκρίνεται αυτή η περιοχή εκεί με μπέρδεψε 1488 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 92 ένδυ. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 18. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 89 εννέα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 1548 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Από κοινού 1549-1550 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1553 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1559 υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1560. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 31 προς 28. Εγκρίνεται. Εγκρίθηκε 1560. 1561. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1563. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1566. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος για το 66. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 29 προς 29. Απορρίφθηκε. Είχατε όμως δίκιο που ζητήσατε έλεγχο. 29, 29. 1784. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1785 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1786 και 105 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεν είναι σαφές έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Πενήντα ένας προς οκτώ. Κανείς δεν σήκωσε το χέρι φαίνεται. Για το 1786 ψηφίζουμε μόνο την προφορική τροπολογία. Σαφές. Όπως. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι απλώς για να διορθώσω κάτι που νομίζω όλες οι ομάδες θα το στηρίξουν. Απλώς το παραβλέψαμε όταν ετοιμάζαμε τις συμβαστικές λύσεις. Το electricity undertakers να αντικατασταθεί από το network operators, φορείς του διαδικτύου. Νομίζω είχαμε συμφωνήσει όταν συζητήσαμε το συμβαστικό πακέτο και εκπανοποιεί όλες τις ομάδες, σε όλες τις συνθήκες. Συμφωνείτε όλοι. Λοιπόν, ψηφίζουμε αυτή την προφορική τροπολογία 1787. Την προφορική τροπολογία μόνο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 1788. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 1789. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 1790 και 91 μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 1792. Έλεγχος για τη 1790 και 91. Άρχεται η ψηφοφορία. Πάλι είναι υπεράριθμα μέλη του ΕΛΚ κατά έναν. Περισσεύει ένας του ΕΛΚ. 28 προς 31. Απορρίπτεται. 1792. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 106. 106 της ΕΝΒ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 1793. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτε. 107 της ένβη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 1796. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 108. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 1797 υπέρ κατά έλεγχος 1797 πέρας 29 προς 30 απορρίπτεται Χολ 1798 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Πέρας και πάλι περισσεύει ένας από το έλεγχο. Okay. 31 a 25. 31 προς 25 εγκρίνεται. 1800 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1809 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 123 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος για την 123. Άρχεται η ψηφοφορία. Πάλι περισσεύει ένα στο ΕΛΚ. Πέρας. 28 προς 30 απορρίπτεται. 124 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 125 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. NV1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 126 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. NV2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 132 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΦΑΜ 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 138 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος για την 138 άρχεται η ψηφοφορία και πάλι περισσεύει ένας του ΕΛΚ πέρας 31 προς 29. Εγκρίνεται. 141 και NV3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 26 προς 32. Απορρίπτεται. 142 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 143 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 144 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 147 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται, πιστεύω. Για την 147. Ένας από το ΕΛΚ περισσεύει. Πέρας. 25 προς 33. Απορρίπτεται. 148 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος. 148. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 33 προς 27 εγκρίνεται. Μπράβο. 149. 149 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 150 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται από τις ομάδες, δεν κατάλαβα όμως με την ανάταση χειρών έλεγχος. Πέρας, 33 προς 26, εγκρίνεται. Εγκρίθηκε 150. 152. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Από κοινού. 155, 156. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος έλεγχος για την 155-156. Πάλι περισσεύει ένας του ΕΛΚ. Ωραία. Πέρας. 26 προς 33. Απορρίπτεται. 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος για την 157. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 29 προς 31. Απορρίπτεται. 159. Χολ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 160. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 161 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έλεγχος για την 161. Πέρας, 31 προς 28. Εγκρίνεται. Τώρα από κοινό, 162 και 163 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 164 υπέρ κατά αποχές απορρίβεται. 166 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 164. 174, συγγνώμη, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 175, υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. 175. Πέρας. 31 προς 29. Εγκρίνεται. Για την 184 τώρα, 184, προφορική τροπολογία, ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 188. Με συγχωρείτε, μπορείτε να μας πείτε τι ψηφίζουμε με την προφορική τροπολογία. Ψηφίζουμε την αρχική τροπολογία που διαγράφει τους όρους or occupied, διότι δεν είναι σαφές για μένα τι ακριβώς ψηφίζουμε. 184. Τσίτσεστερ. ψηφίζουμε την τροπολογία Τσίτσεστερ μαζί με την προφορική της τροπολογία, δηλαδή με την προστίκη της προφορικής. Η προφορική τροπολογία δηλαδή είναι να διαγραφούν οι όροι or occupied. Ναι, διαγράφονται αυτοί οι όροι με την προφορική τροπολογία. Μα ψηφίσαμε. 184 ψηφίσαμε. Μπορούμε να ψηφίσουμε ξανά για να είμαστε βέβαιοι. Μάλιστα. 184 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Πέρας. 30 προς 28. Εγκρίνεται. Εκατόν ογδόντα οκτώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 183. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 181 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 185 και NV5 από κοινού υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 190 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θαμ 2 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έλεγχος για το ΦΑΜ2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 24 προς 33 απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 200 υπέρ. Εκατόν ενενήντα Με συγχωρείτε. Εκατόν ενενήντα εννέα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Συγκεχημένη κάπως η ψηφοφορία στο αποτελεσμά της. Έλεγχο να κάνουμε. 199. Πέρας της πληροφορίας 32 προς 26. Εγκρίνεται. 201 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 205 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 208 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. ΘΑΜ 4 επόμενη σελίδα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 214 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος για τη 214. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 42 υπέρ, 15 κατά. Εγκρίνεται. 221 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 223 υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρι... Απορρίπτεται. 7. Υπέρ. Όχι, καταπίπτει. 3. Τροπολογία 3. Όχι, 217. 217 τσίτσεστερ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τρία Υπέρ. Ο κύριος Τούρμες. You check again. Μπορείτε σας παρακαλώ να ελέγξετε και πάλι αν καταπίπτει η επτά του περιβάλλοντος. Γιατί δεν εγκρίθηκαν οι δύο προηγούμενες τροπολογίες ή μήπως φάλω. Όχι, όχι, συγγνώμη, εγώ έκανα λάθος, λέει ο κύριος Τούρμας. Scusi, siamo l'emendamento 3. Τροπολογία 3 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 231. Όχι. 231 την ξεχνάμε. 232, 233 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 238 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 200 όχι καθόλου 236 236 και 37 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 241 υπέρ κατά αποχές μοιάζει να απορρίπτεται. 242 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 243 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Όχι, έλεγχος. 243 έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 28 προς 31. Απορρίβεται. 244. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 256. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 252. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 248 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 257 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 258 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 262 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 264, 65 και 66 από κοινού. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 267 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 268 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 200 ελέγχουμε για τη 268. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 35 προς 21. 268 εγκρίνεται λοιπόν. 269 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ένβη 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 263. 273, συγγνώμη, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 274. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 276. Υπέρ. 274. Κάνουμε έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 28 προς 30. 274 απορρίπτεται. 276 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 277 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 278 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 279 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 280 και NV10 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Φάν 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Ένβι 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 281 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Έλεγχος για το 281. Πέρας. Παναγιά μου, 47 προς 13. Συγχαρητήρια, πολύ ωραία. 282. 280, ή 281 εγκρίθηκε. 282. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται.

υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 286 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 287 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 12, Έντι 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. ΘΑΜ 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Όχι, όχι, με συγχωρείτε. ΘΑΜ 7 έλεγχος. Εγώ νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ας ελέγξουμε. Πέρα. 16 προς 42. Απορρίφθηκε. ΕΝΒΙ 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 302 υπέρ ναι 302 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος. Κιούζα. Πέρας. 32 προς 28. Εγκρίνεται. NV19. NV19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. NV21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 306 υπέρ κατά αποχές έλεγχος 306 Πέρας 28 προς 30 απορρίπτεται. Απορρίφθηκε. 122. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 121. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ξεχάσαμε μία τροπολογία. Ξεχάσαμε μία τροπολογία στη σελίδα 100 πάνω κάτω της κυρίας Φόρντ. Ήταν η τροπολογία 1489. Άρθρο 17, παράγραφος 2. Σελίδα 97. Για τους σοσιαλιστές ή 100 για το ΕΛΚ. Δεν είμαι βέβαιη. Άρθρο 17, παράγραφος 2, σελίδα πάνω κάτω 198, 100, κάτι τέτοιο. Τροπολογία 1489 της κυρίας Φόρντ, η οποία δεν ψηφίστηκε. Τη βρήκατε όλοι. Ας ψηφίσουμε λοιπόν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Ωραία. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 51 υπέρ, 6 κατά, 3 αποχές. Και τώρα ψηφοφορία για την έναρξη διαθεσμικών διαπραγματεύσεων, δηλαδή με το Συμβούλιο, ψηφίζουμε αμέσως, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 31 υπέρ, 22 κατά, 5 αποχές. Θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Questo qui è del GPL, mm. io eh, Piriglia.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 Αρχίζουμε αμέσως την ψηφοφορία για την έκθεση Κάριν. Σας παρακαλώ να καθίσετε. Έχουμε ακόμη και άλλη έκθεση να ψηφίσουμε. Σας παρακαλώ όλοι να καθίσετε. Διότι έχουμε και άλλη ψηφοφορία. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ξεκινούμε, Ξεκινάμε με... με την έκθεση Κάριν με τη συμβιβαστική ένα Έκθεση Κάρινς. Όποιος δεν ενδιαφέρεται παρακαλώ πάρα πολύ να εγκαταλείψει την αίθουσα άμεσα. διότι πρέπει να συνεχίσουμε τις ψηφοφορίες. Όποιος δεν θέλει ας εγκαταλείψει την έκθεση την αίθουσα. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 1 τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, μαζί 10, 61, 62 και 11 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι απερίφθη, αλλά θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο γιατί υπάρχει μεγάλη σύγχυση. Ξεκινά ο ηλεκτρονικός έλεγχος για την 10, 61, 62 και 11. Κάποιος άλλος ε, ψηφίζει ακόμη. Τελειώσαμε. 27 υπέρ, 21 κατά. Τροπολογία 60 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 63 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ, κατά, αποχές Εβδομήντα. Ηλεκτρονικός έλεγχος ξεκινά. Λίγοι. 18 υπέρ, 31 κατά. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται μαζί 14 και 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, το 75 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές 97 πρώτο μέρος ηλεκτρονικός έλεγχος ξεκινάει. Λίγη. 23 υπέρ 29 κατά απερίφθη. 110 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 112 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 113 και 13 ίντα ε, μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 114 και 16 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 16 και 115 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 121 και 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 122 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 124 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 124. Λίγη. 24 υπέρ, 30 κατά, περίφθη. 125 υπέρ με συγχωρείτε πριν από αυτήν είναι η τροπολογία 20 τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 126, 21 και 17 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 131 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η συμβεστή 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το 24. Ε, Ξεκινά για το πρώτο μέρος του 24, της τροπολογίας 24. 28 υπέρ, 26 κατά, ενεκρίθη. Τροπολογία 2 μαζί με την 29, 30 και 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι ενεκρίθη, αλλά κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Ε, ανοίγει, ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγοι. 33 υπέρ, 22 κατά, είναι κρίθη. 27 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά 2 τη ΣΥΝΤΑ. υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 33. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 34. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 3. Ίντα. Υπέρ, Η γραμματεία λέει ότι πρέπει να την ψηφίσουμε διότι η, η τροπολογία 3 λοιπόν υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 3 λίγοι. Απερίφθη 20 υπέρ και 33 κατά. 35 υπέρ. Κατά αποχές ενεκρίθη. 36 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. 37 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. 38 και 39 υπέρ κατά α, και 40 με συγχωρείτε υπέρ κατά αποχές απερίφθη 41 και 43 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 42 μάλλον 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για τις 48 Κιούζο, Πέρας. 28 υπέρ, 18 κατά. 49 υπέρ. Κατά. Απερίφθη. 6 υπέρ. Κατά αποχές ενεκρίθη. 50 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 51 υπέρ κατά αποχές ενεκρίθη. 53 και 5 μαζί υπέρ. Με συγχωρείτε, πρώτα το 7, ξεχάσαμε το 7, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνουμε. 53 και 5 μαζί υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 και 6 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 και 7 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ ε, κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έλεγχος για τη, ηλεκτρονικός για την τροπολογία 9 ξεκινά λίγη 25 υπέρ 28 κατά απερίφθη τελική ψηφοφορία ξεκινά η ψηφοφορία ξεκινά η τελική ψηφοφορία όπως είπαμε Λίγοι. 48 υπέρ και πέντε κατά. Συγχαίρουμε. Και τώρα ψηφίζουμε για τις ε, θεσμικές ε, διαπραγματεύσουμε το Συμβούλιο. Ξεκινάει η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Λίγη. Σαράντα υπέρ και τέσσερις κατά. Ε, υπομονή έχουμε ακόμη δύο ψηφοφορίες οπότε υπομονή στα γρήγορα περνάμε στην τελική ψηφοφορία για το, την έκθεση Γκέρεκ άρθρο 44 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 48 επαναλαμβάνω υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 και 50 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Λίγοι. 28 υπέρ εγκρίθηκε. 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 μόνο το δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 75. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 78. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 79. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 80. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 81. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 88 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 89 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 90 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 91 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 92 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 93 υπέρ, κατά, έλεγχος. Sul 93 stiamo 93 ψηφίζουμε. Votazione chiusa. Πέρας. Εψήφισαν άπαντες, εγκρίνεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά Αποχέ. εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά Αποχέ. εγκρίνεται. 1 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά Αποχέ. εγκρίνεται. 36 υπέρ κατά Αποχέ. εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. 38 37 έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 24 προς 23. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. 37. 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν ξέρω αν είναι όπως πριν. Ας ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. 38. Πέρας. 25 προς 21. Εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά, απόχέ εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά, απόχέ, εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. 7 υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. 8 υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. 40 υπέρ, κατά, απόχέ απορρίπτεται. 41 υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Ναι, με συγχωρείτε, πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά ούτω ή άλλω. Μπερδεύτηκα. Ανοιχτή ψηφοφορία ονομαστική για την έκθεση. Πέρας. ...38 υπέρ 5 κατά 2 εποχές εγκρίθηκε. Τελευταία ψηφοφορία για σήμερα το πρωί. Έκθεση Τζαβέλα. Παράγραφο 1. Τροπολογία 1. Υπέρ. Ψηφίζουμε την έκθεση Τζαβέλα.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 με την προφορική τροπολογία κατά αποχέ, εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία Ψηφίζουμε ηλεκτρονικώς. E voto chiusa.